Αγαπητοί συνάδελφοι, να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Στην ε, ημερήσια διάταξη έχουμε δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ατζέντα για τις νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας. Να δώσουμε απευθείας το λόγο στον Επίτροπο Άντορ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Σήμερα έχουμε στην Ευρώπη 23 εκατομμύρια ανέργους που σημαίνει περίπου το 10% ε, του ενεργού πληθυσμού είναι ο δείκτης της ανεργίας. Η κατάσταση αυτή ανέκυψε ως αποτέλεσμα και συνέπεια της χρηματοοικονομικής κρίσης. Και πραγματικά ε, φοβούμαστε δραματικές συνέπειες. Αυτή η κατάσταση όμως δεν απέτρεψε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το να προτείνει στη στρατηγική του 2020 φιλόδοξου στόχους. Και όντω είναι φιλόδοξοι οι ε, στόχοι μας και μάλιστα ε, μέσω πρόθεσμη. Μέχρι το 2020 θέλουμε να απασχολείται το 75% του πληθυσμού ανδρών και γυναικών. Και άλλος στόχος είναι ε, πλέον και μια ατζέντα για τις νέες δεξιότητες και θέσεις ε, εργασίας. Να σας εξηγήσω πώς θα προχωρήσουμε. Αυτό είναι ε, συμπροματικό με την πρωτοβουλία νεολαία σε κίνηση για τους στόχους στην ανάπτυξη, στην απασχόληση. Βεβαίως η κρίση ε, οδήγησε σε απώλεια εκατομμυρίων θέσεων εργασίας και έχουμε και τεράστιο διεθνή ανταγωνισμό. Αλλά αυτός δεν είναι λόγος να διστάζουμε να λάβουμε δράση. Το αντίθετο, θα πρέπει να ε, διαμορφώσουμε καλύτερα το μέλλον μας με καλύτερες θέσεις εργασίας και περισσότερες και αυτό είναι στα χέρια μας. Ε, είναι σε μεγάλο βαθμό η πολιτική απασχόληση μεν, υπόθεση των κρατών μελών, αλλά επειδή χαράζουμε και εμείς πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κοινωνική Εταιρεία θα πρέπει να κάνουμε και εκείνο που μας αναλογεί να επιτρέψουμε στους εργαζομένους να ε, προχωρήσουν νέες ιδέες και δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Η νέα γενιά να υποφεληθεί από το κοινωνικό μοντέλο που έχουμε αναπτύξει στην Ευρώπη. Για όλους τους εργαζομένους χρειαζόμαστε καλύτερες συνθήκες εργασίας και μεγαλύτερη ποιότητα εργασίας. Η ατζέντα για τις νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας ορίζει τέσσερις τομείς. λειτουργία της αγοράς εργασίας, δεξιότητες, ποιότητες εργασίας και ε, συνθήκες εργασίας και δημιουργία θέσεων απασχόληση. 13 είναι οι δράσει συγκεκριμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, σε συνεργασία με κυβερνήσει, κοινωνικού εταίρους και κοινωνία των πολιτών. Καταρχάς θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι λειτουργεί καλύτερα η αγορά εργασία με μεταρρύθμιση στην αγορά έτσι ώστε να υπάρχει απαραίτητη ευελιξία και να συνοδεύεται από την απαραίτητη ασφάλεια. Τα τελευταία δύο χρόνια μάθαμε ότι οι πολιτικές ευελιξίας με ασφάλεια ε, security, βοήθησαν. Τώρα θα πρέπει να συζητήσουμε όλα τα στοιχεία της πολιτικής αυτής με τα κράτη-μέλη και πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε για να έχουμε ε, μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση για ευελιξία με ασφάλεια. Να ε, υπάρχουν ε, συνθήκες εργασίας ευέλικτες μεν, αλλά στις οποίες θα μπορούμε να βασιζόμαστε με εκπαίδευση και σωστές θέσεις απασχόλησης. Στην Ευρώπη αυτό ποικίλει πάρα πολύ. Υπάρχουν συλλογικέ συμβάσει ενώ ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο εργασία με τις ίδιες συνθήκε και ε, την ίδια απασχόληση έχουμε εργαζομένους με επισφάλεια, με ε, χαμηλή προστασία και αβέβαιες ε, συμβάσει περιορισμένου χρόνου. Ένας τρόπος επίλυσης αυτό είναι η ατζέντα για τις νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας για να διευρυθεί ε, η σύμβαση αορίστου χρόνου και να καλύπτει και τη διαβίου μάθηση και τη μετεκπαίδευση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό όλων των εργαζομένων. Αυτό θα ε, βοηθήσει τους εργαζομένους να έχουν πλήρη δικαιώματα με αρκετή ευελιξία αλλά συνεχώς μειούμενη κατά τη διάρκεια της άσκησης. Πολλές φορές διστάζουν ε, να προσλαμβάνουν οι ε, επιχειρηματίε ασκουμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίση είναι νέε δεξιότητε και για την αγορά και για το μέλλον. Γνωρίζουμε ότι ήδη από τώρα ορισμένοι εργοδότε, δεν μπορούν να καλύψουν τι θέσει απασχόληση γιατί δεν βρίσκουν του εργαζόμενου με τα απαραίτητα προσόντα και τι δεξιότητε. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει ότι χρειαζόμαστε περισσότερε δεξιότητε, αλλά και τι σωστέ δεξιότητε, αλλά και ε, έχουμε κάποια ε, ασυνέχεια η ε, απόκληση της εκπαίδευσης στην Ευρώπη από τις ανάγκες ε, των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Ασκούμενοι γιατροί, δικηγόροι, νοσηλευτές και άλλοι χρειάζονται περισσότερο, ακόμα και πρόσωπα που θα απασχολούνται στην πράσινη οικονομία. Χρειάζονται τακτικά εργαλεία, λοιπόν, για μεγαλύτερη διαφάνεια για τις ανάγκες που έχουμε στις δεξιότητες, για καλύτερη συσχέτιση ε, της εκπαίδευσης με την εργασία, με ένα πανόραμα για να καταλάβουν και ε, οι εργαζόμενοι και οι υποψήφοι εργαζόμενοι τι δεξιότητες χρειάζονται στο μέλλον. Η κυρία Βασιλείου θα επεκταθεί περισσότερο σε αυτό το θέμα. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους τους ενδιαφερομένους για να καλυφθεί το χάσμα εκπαίδευσης, κατάρτισης και ε, αγοράς εργασίας. Στη συνέχεια, προτείνουμε να βελτιωθεί η ποιότητα των θέσεων ε, εργασία με καλύτερε συνθήκες εργασία. Είναι πάρα πολύ φιλόδοξη η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και τώρα καλείται να αναθεωρηθεί. Η ε, εφαρμογή στην πράξη μας διδάσκει και μας δείχνει πού και πώς ε, χωράει η βελτίωση. Για να, λειτουργεί καλύτερα η νομοθεσία θα πρέπει να εγγράφεται στη νέα τεχνολογία, στη νέα σχήματα απασχόλησης, να είναι εύληπτη και εύκολα ε, όλα αυτά στην εφαρμογή τους για τους εργοδότες και για τους εργαζομένους. Οδηγία για το ωράριο εργασίας θα πρέπει να εφαρμόζεται σωστά για να βελτιώνεται επίσης και η εφαρμογή τη απόσπαση των εργαζομένων τη αντίστοιχη οδηγία και ε, πάντα με σεβασμό στην ασφάλεια και την υγιεινή. Για την αναθεώρηση λοιπόν η ατζέντα προτείνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει λεγόμενα ήπια μέσα από κώδικες συμπεριφοράς και συστάσεις μέχρι ε, καθοδήγηση για την εφαρμογή, ανταλλαγή καλόπρακτικών, συγκριτική αξιολόγηση. Προσβλέπω στη συζήτηση μαζί σα και είμαι πεπισμένο ότι μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη-μέλη και τους κοινωνικού εταίρους μπορούμε να κάνουμε την εργασία καλύτερη. Βεβαίω χρειάζεται να δημιουργήσουμε και περισσότερε θέσει εργασία, για την ανάπτυξη, αλλά είναι ακόμα πάρα πολλά τα εμπόδια που ορθώνονται στο δρόμο μας. Προτείνουμε να βελτιωθούν οι συνθήκες πλαίσιο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε τομείς που κινούνται γρήγορα στην έρευνα και στην ανάπτυξη με μείωση του γραφειοκρατικού ε, φόρτου, με μείωση της φορολόγηση εργασίας και βοήθεια προς τους εργοδότες. Προτείνουμε και δράση για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και να βοηθήσουμε, να υποστηρίζουμε εκείνους που ξεκινούν μια επιχείρηση ε, ή μόλις ε, πρόσφατα ξεκίνησαν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε το νέο μικρό χρηματοδοτικό μέσο ακριβώς για να μπορούν να ε, δημιουργούν ε, οι ενδιαφερόμενοι επιχειρήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρα πολλά ταλέντα, αλλά θα πρέπει οι ιδέες, οι καινοτομίες να οδηγούν και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε τι προτεραιότητε για το πώ θα προοδεύσουμε προ την πλήρη απασχόληση. Ατζέντα για νέε δεξιότητε και θέσει εργασία μπορεί να βοηθήσει αυτή μόνο εφόσον συνεργαστούμε όλοι. Απευθύνω έκκληση προ όλου να παίξει ο καθένα το ρόλο του στην προσπάθειά μα αυτή να φτάσουμε στην πλήρη απασχόληση στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο Άντορ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στην Επίτροπο Βασίλη. Βασιλείου για να κάνει και τη δική της παρουσίαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που παρουσιάζουμε από κοινού με τον Επίτροπο Άντορ τη νέα σημαντική πρωτοβουλία, μια ατζέντα, ένα πρόγραμμα εργασιών για νέε δεξιότητε και θέσει εργασία. Καλύτερη παιδεία και κατάρτιση θεμελιώδεις στόχοι για να εφοδιάσουμε τους εργαζόμενους με τις, προσ... με τις δεξιότητες και τα προσόντα που χρειάζονται για να βρουν μια δουλειά, να παραμείνουν σε αυτή και να προετοιμαστούν για τις μελλοντικές θέσεις εργασίας. Γι' αυτό και θα πρέπει να επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό και στην ικανότητα του κόσμου να καινοτομεί, να δημιουργεί νέες επιχειρήσεις και νέες θέσεις απασχόλησης. Χωρίς ε, σημαντική και διαρκή επένδυση σε υψηλά επίπεδα δεξιοτήτων και σε παιδεία θα, δεν θα μπορέσουμε να βγούμε γρήγορα από την κρίση. Οι δεξιότητε και τα προσόντα βρίσκονται στην καρδιά τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 2020 για ευφυή e e, αηφόρα ανάπτυξη που δεν θα περιθωριοποιεί κανένα. Γι' αυτό και έχουμε δύο σημαντικέ πρωτοβουλίε, την νεολαία σε κίνηση και το πρόγραμμα εργασιών για νέες δεξιότητες και εργασίες με, με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδεία, την κατάρτιση αλλά και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Σήμερα με την πρωτοβουλία αυτή θέλουμε να προβληματιστούμε πώς η παιδεία και η κατάρτιση θα συμβάλλουν στο να υλοποιήσουμε το στόχο μας για 75% ποσοστό απασχόλησης μέχρι το 2020. Γιατί θα έχουμε 16 εκατομμύρια νέες θέσεις απασχόλησης μέχρι το 2020 με ήδη υψηλά ειδικευμένους. Ενώ η μείωση των ανειδίκευτων θέσεων θα είναι γύρω στα 12 εκατομμύρια. Έχουμε πάνω από 8 εκατομμύρια ε, άνεργους στην Ευρώπη που δεν έχουν σημαντικές ε, δεξιότητες. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της παιδείας της επιμόρφωσης. Επίσης να αναγνωρίσουμε τη διαβίου κατάρτιση ως νευραλγικό πυλώνα της στρατηγικής για την ευελιξία και την ασφάλεια, ώστε η αγορά εργασίας μας να λειτουργεί πιο εύρυθμα, όπως τόνισε και ο Επιτροπός Άντορ. Συμφωνούμε όλοι ως προς τη διάγνωση. Οι δεξιότητες, τα προσόντα μπορούν να, να εξασφαλίσουν και να βελτιώσουν την α, κινητικότητα στην αγορά εργασίας. Η διαβίωση όμως κατάρτιση δυστυχώς δεν αποτελεί πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων δεν θα πρέπει να είναι πολυτέλεια μόνο για του υψηλά ειδικευμένους. Είναι αναγκαιότητα για όλους. Και οι ανειδίκευτοι θα έχουν ελάχιστες ευκαιρίες να συμμετέχουν σε διαβίου κατάρτιση σε όλα τα κράτη-μέλη. Μέχρι στιγμή αυτό συνέβαινε, αλλά αυτό θα πρέπει να αλλάξει με κοινέ προσπάθειε όλων των εταίρων, των κυβερνήσεων, των εργοδοτών και των ε, επιχειρήσεων. Θα πρέπει να εφοδιάσουμε του εργαζόμενου με τι απαραίτητε δεξιότητε και τι σωστέ δεξιότητε. Δεν θα πρέπει να αναβαθμίσουμε τι δεξιότητε των ίδιων εργαζομένων όσων βρίσκονται στην αγορά εργασία, αλλά να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα να έχουν από την αρχή οι πολίτε το σωστό μείγμα εφοδίων και προσόντων ώστε να προσαρμόζονται σε μια συνεχώ μεταβαλλόμενη κοινωνία και αγορά εργασία. Επίση, θα πρέπει να εστιαστούμε καλύτερα στι απαραίτητε δεξιότητε στην αγορά εργασία και με αυτή την προοπτική θα υποβάλουμε νέο πανόραμα, ένα νέο τοπίο των ευρωπαϊκών δεξιοτήτων που θα μας κατατοπίζει όχι μόνο για το τι δεξιότητες απαιτούν οι εργοδότες, αλλά θα επικεντρωθούμε και στις δεξιότητες που θα καταστούν απαραίτητες στο μέλλον για να προετοιμάσουμε τους νέους μας να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, να προσαρμοστούν και να εργάζονται σε θέσεις απασχόλησης που σήμερα μπορεί να μην υπάρχουν ακόμη, θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε εκπαιδευτικά συστήματα που θα εξασφαλίζουν το σωστό μείγμα δεξιοτήτων. Θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στις στοιχειώδεις δεξιότητες, ανάγνωση, μαθηματικά, θετικές επιστήμες, γιατί είναι πολύ σημαντικό να, καταποτε... να καταπολεμήσουμε ε, την ε, πρόορια εγκατάλειψη της εκπαίδευσης ή τις χαμηλές επιδόσεις στα σχολεία. Γι' αυτό από τον Ιανουάριο θα συγκροτήσουμε μία ομάδα υψηλού επίπεδου για τον αλφαβητισμό. Θέλουμε μια κοινωνία που θα στηρίζεται στη γνώση. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε παιδιά που θα έχουν καλύτερε επιδόσει στα μαθηματικά, στι επιστήμες και στην τεχνολογία. Βέβαια, θα πρέπει να εστιάσουμε τι προσπάθειέ μα και στην απόκτηση κάποιων εγκάρσιων προσόντων και δεξιοτήτων, που είναι σημαντικά για την απασχολησιμότητα, όπω εκμάθηση ξένων γλωσσών, ε, ψηφιακός αλφαβητισμός και δεξιότητες ως προς την ανάληψη πρωτοβουλειών. Επίσης ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που θα απαιτηθούν από τις μελλοντικέ ε, εργασίες. Για παράδειγμα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις, ε, στις φιλοπεριβαλλοντικά κτίρια, στα στην υγεία, στις ευφυείς συγκοινωνίες. Ακόμη και σε περιόδους κρίσης με υψηλή ανεργία, ορισμένοι εργοδότες εξακολουθούν να έχουν προβλήματα στις προσλήψεις. Γι' αυτό με το πρόγραμμά μας θέλουμε να συνδεριάσουμε καλύτερα τα προσόντα με τις ε, δυνατότητες και ευκαιρίες ε, απασχόλησης. Γι' αυτό και προτείνω ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων που θα επιτρέπει στους πολίτες να καταγράφουν το προσόντα τους με σαφή και συγκρίσιμο τρόπο. Και μάλιστα θα οδηγηθούμε σε ένα πολύ δημοφιλές ε, ε, ευρωπαϊκό διαβατήριο και ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να βρούμε το σωστό μείγμα δεξιοτήτων και να αναζητήσουμε νέες μορφές συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς κύκλους, με τους εργοδότες, τι επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους όπω τα συνδικάτα και ε, δημόσιες υπηρεσίες απασχόληση και εργασία. Αγαπητοί συνάδελφοι και ευρωβουλευτέ, με την στρατηγική του 2020 θέσαμε του στόχου μα και τι προσδοκίε μα, Είναι η ώρα να σημειώσουμε πρόοδο προς την υλοποίηση αυτών των προσδοκιών και στόχων και να επαναπροσδιορίσουμε τη στρατηγική μας για τις μεταρρυθμίσεις. Η ατζέντα για τις νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας εξηγεί το πώς θα συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι. Για να εξέλθουμε από την κρίση θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια ανταγωνιστική οικονομία που θα στηρίζεται στη γνώση και που θα προσφέρει περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Επίτροπο. Να δώσουμε τώρα το λόγο στους αγορητές, οι οποίοι θα μιλήσουν εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, ξεκινώντας από τον κύριο Ορή για 1,5 λεπτό. Ε, ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρία Επίτροπε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει κατά παράδοση τους επιτρόπους, μερικές φορές βέβαια τους ε, ασκεί κριτική. Αυτή τη φορά όμως είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο από αυτά που, ακούσαμε και από τους δύο επιτρόπους και τον κύριο Άντορ και την κυρία Βασιλείου. Χάρη και για τους ορισμούς ε, που μας παρουσιάσατε, για τους στόχους που μας ε, παρουσιάσατε. Τέσσερι προτεραιότητε. Καλύτερη αγορά εργασία, καλύτερε θέσει εργασία με περισσότερε δεξιότητε, καλύτερε πολιτικέ και καλύτερε συνθήκε εργασία. Είμαι υπέρ όλων αυτών των στόχων και βέβαια θα είναι δύσκολο να τους εφαρμόσουμε, αλλά συμφωνώ με αυτά που είπατε και για το flex security, την ευελιξία με ασφάλεια. Θα πρέπει όμως επιτέλους να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες, γιατί πολύ συχνά χρησιμοποιούμε αυτή την έννοια του flex security, αλλά ίσως δεν την ερμηνεύουμε με τον ίδιο τρόπο. Επίσης πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να αντιδράσουμε με σωστό τρόπο προς τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην αγορά εργασίας και στους χώρους εργασίας, αλλά η οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων δεν θα πρέπει να αντικατασταθεί από μια νέα οδηγία. Συζητούμε προβλήμα προβλήματα εφαρμογής και τις αδυναμίες και κάποιες προσαρμογές που θα χρειαστούν. Αλλά οι ατυπικές μορφές εργασίας είναι επίσης σημαντικό θέμα, γιατί θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτή τη νέα κατάσταση και από άποψη κοινωνικών εισφορών και κοινωνικής ασφάλειας. Θα πρέπει να προωθήσουμε φυσικά την κινητικότητα, να συνεργαστούμε και με τις αρμόδιες κρατικές αρχές. Βλέπω ότι ο πρόεδρος ε, με προειδοποιεί για την εξάντληση του χρόνου μου και σίγουρα δεν ε, θέλουμε ανειδίκευτους μόνο εργαζομένους και σίγουρα θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την ανεργία. Θα πρέπει να βοηθήσουμε και του ανειδίκευτου να βελτιώσουν τι δεξιότητε και τα προσόντα με περισσότερη κατάρτιση. Η κυρία Συμβάλα Λάπτη για 1,5 λεπτό τώρα. Ε, άκουσα με πάρα πολύ χαρά τις εισηγήσεις των δύο επιτρόπων. Σε καιρό κρίσης και μάλιστα έντονης έχουμε ανάγκη από το όραμα. Οι δύο εισηγήσεις μας προσέφεραν ένα όραμα. Είναι φιλόδοξες έδωσαν τέσσερις στόχους τους οποίους νομίζω ότι κάθε ευρωπαίος πολίτης θέλει να υποστηρίξει αλλά πάντα σε όλα τα ωραία υπάρχει και ένα αλλά. θέλω να επισημάνω πρώτον το θέμα της ασφάλειας. η ευελιξία με την ασφάλεια πρέπει να πηγαίνουν χέρι χέρι και η γνώμη μας είναι ότι προτεραιότητα πρέπει να την έχει η ασφάλεια το θέμα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι πάρα πολύ βασικό διότι όπως πολύ σωστά επεσήμανε ο επίτροπος andor έχουμε ανάγκη όχι μόνο νέες δεξιότητες αλλά και τις παλαιές δεξιότητες να τις καθοδηγήσουμε εκεί που πρέπει. υπάρχουν τα ζητήματα της επιχειρηματικότητας πρέπει να διευκολυνθούν οι νέοι να μπορούν να ανοίξουν τη δική τους δουλειά πρέπει να διευκολυνθούν οι επιχειρηματίες να μπορούν να προσλαμβάνουν περισσότερο. και κλείνοντας αναφέρομαι σε αυτό το πολύ ωραίο που είπε η επίτροπος βασιλείου ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο για τις δεξιότητες. εκεί όμως αμέσως έρχεται το μυαλό μου στους αποσπασμένους εργαζόμενους και σκέφτομαι και ρωτώ και τελειώνω κύριε πρόεδρε αμέσως εάν εγώ έχω ένα διαβατήριο με εξαιρετικές δεξιότητες και προέρχομαι από μια χώρα α και πάω να εργαστώ σε μια χώρα β θα έχω λυμένο το θέμα των εργασιακών μου σχέσεων θα είμαστε στο πλευρό σας θα παρακολουθούμε και θα αγωνιζόμαστε μαζί σας. ευχαριστώ. Ε, Συνάδελφοι, σας παρακαλώ να τηρείτε λίγο τους χρόνους, διότι έχουμε καθυστερήσει αρκετά από τον προβλεπόμενο χρόνο μας. Η κυρία Μαρία Χάρκιν για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε ε, Επίτροπη, ε, θα αναφερθώ σε μία από τις τέσσερις προτεραιότητες. Περισσότερες πολιτικές για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση και τη ζήτηση. Σύμφωνα με το έγγραφο θα πρέπει να έχουμε περισσότερες θέσεις απασχόλησης, ναι, δημιουργία, αλλά ε, είναι τεράστια η κρίση ε, στην Ευρώπη. Εγώ που είμαι προβουλευτής από την Ιρλανδία ξέρω πολύ καλά ε, πώς μας καλούν τώρα να επιβάλλουμε μέτρα λιτότητας και φοβάμαι ότι θα περιορίσει κάθε δυνατότητά μας αυτό. Ερωτώ, αυτή η ατζέντα για νέες θέσεις εργασίας δεν αφορά την Ιρλανδία ή την Ελλάδα ή όποια χώρα είναι στο μνημόνιο. Και πού θα βρεθεί η ανάπτυξη και πού θα βρεθούν οι θέσεις εργασίας. Είναι εξαιρετικέ οι ιδέες του εγγράφου, εγώ δεν προσπαθώ να το υποτιμήσω, αλλά ε, είναι κρίσιμο να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε επενδύσεις, έρευνα, ανάπτυξη και πώς θα το συνδέσουμε στο σύστημα παραγωγής. Είναι απολύτω απαραίτητο αυτό. Κοινωνική οικονομία, ε, ε, μικρό επιχειρήσεις, εταιρείε αλληλοβοήθειας, όλα αυτά καλά σε τοπικό επίπεδο είναι πολύ επίκαιρα και ε, πιστεύω ότι πραγματικά η τοπική κινητοποίηση είναι πολύ σωστή ε, και οι επιχειρήσεις αλλοβοήθειας που δεν είναι και κερδοσκοπικές μπορούν να βοηθήσουν για την ανάπτυξη. Η πρόθεση της επιχειρηματικότητας θα επιτρέψει στους πολίτες τους ίδιους να παίξουν ένα ε, ρόλο σημαντικό στην ανάκαμψη της οικονομίας και επίση είναι καλό να συνδέουμε τι δεξιότητε με τι θέσει εργασία. Ανησυχώ πολύ. Την περασμένη εβδομάδα ε, ε, είχα μία συνάντηση ε, στο Κοινοβούλιο για την ψυχική υγεία και την ανάπτυξη. Και βγήκε μια Αυστριακή συνάδελφο και είπε σταματήστε να μιλάτε για θέσει απασχόληση και ανάπτυξη. Κανεί δεν σα πιστεύει. Συγκλονίστηκα. Δεν ξέρω πώ κυριαρχεί αυτή η αίσθηση και πώ μεταδίδεται. Πάντω μεταδίδεται. Είναι επίγουσα η κατάσταση και θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουμε νοοτροπία και μυαλά. Ναι, ωραίε οι πράσινε θέσει απασχόληση, αλλά κυρίω οι θέσει απασχόληση επιτόπου και μάλιστα μη κερδοσκοπικέ. Όχι ω υποκατάστατο, αλλά ω αντίβαρο στο κέρδο που έχει κατακλείσει την αγορά και τώρα ε, ε, απειλεί και τη σταθερότητα τη Ένωση και το ευρώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ερίζα Μπετσουρέντερ έχει το λόγο για 1,5 λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε αξιότιμοι κύριοι επίτροποι. περιμένω τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μεγάλες προσδοκίες πρέπει να σας πω για μια νέα όθηση για τους εργαζομένους στην Ευρώπη για να προετοιμαστούν για την οικολογική αλλαγή μια που και ω Κοινοβούλιο για τις πράσινες θέσεις απασχόλησης είχαμε ήδη αναπτύξει πολλές ιδέες, περιμέναμε όντω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τις υιοθετήσει, να τις μεταξελίξει και να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα. Πώς θα γίνει με την οικολογική αλλαγή να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης ή τι υπάρχουσε να τι αξιοποιήσουμε έτσι με τέτοιε δεξιότητε και προσόντα ώστε να διατηρούνται, να μην μπορούν να καταργηθούν. Και να γίνει πιο πράσινη ολόκληρη οικονομία, η βιομηχανία στην Ευρώπη και προ όφελο των εργαζομένων, ανδρών και γυναικών. Ανταυτού εσεί τι κάνετε. Ε, μας παραπέμπετε και ξαναζεσταίνετε το παλιό θέμα flexicurity. Ευελιξία με ασφάλεια. Έτσι θα δημιουργήσουμε νέε θέσει απασχόληση με απορρίθμιση. Μα μόλι τώρα δεν διαπιστώσαμε ότι στην κρίση ακριβώ οι επισφαλεί θέσει απασχόληση είναι τα πρώτα θύματα το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι πλανάστε. Αν νομίζετε ότι μια οικονομία που βασίζεται στη γνώση μπορεί να εδράζεται ε, σε επισφάλεια και ανασφάλεια. Ποντάρετε στη φτώχεια μέσω της εργασίας, αντί να έχουμε εργασία για την ευημερία των πολιτών. Η φτώχεια είναι κακό συνοδός της πρόοδου θέλουμε μια οικολογική αλλαγή, ε, μια επιθετική ε, στάση ε, προς την οικονομία και ιδιαίτερα για τους χαμηλόμισθους. Παρακαλώ, χρειάζεται νέες δεξιότητες και η δική σας δήλωση. Να μην παραμείνετε σε αυτό το τόσο χαμηλό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μίλαν Κάμπρος νομίζω ότι απουσιάζει. Να περάσουμε τότε στην κυρία Μάρα Μπιτζότο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η παρέμβασή μου δεν θα ήθελα να είναι η συνήθι ρητορική. Θα ήθελα μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα εστιάζει περισσότερο στο περιεχόμενο και όχι στον περιέκτη. Θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Η στρατηγική τη Λισαβόνα ε, ε οδήγησε σε ένα νέο σλόγγαν, την Ευρώπη του 2020, αλλά δεν δώσαμε απαντήσει. Τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν. 9,6 ανεργία, 20,2% η ανεργία των νέων. Στην Ιταλία, ένας από τους μεγαλύτερους στον ε, προπολογισμό. Η Ιταλία βρίσκεται σε πολύ ε, κακή κατάσταση και έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό νέων ανέργων. Θα πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικές επενδύσεις ώστε να ετοιμάσουμε επαγγελματίε για τον τομέα της εσωτερικής αγοράς ε, όπου υπάρχουν συγκεκριμένες δυνατότητες θέσεων εργασίας. Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να σημειώσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε διαβίου κατάρτιση. Ο ο κόσμος της βιοτεχνίας δίνει δυνατότητες θέσεις απασχόλησης και μια μοναδική κληρονομιά και θα πρέπει να αναλάβει τα καθήκοντα να υποστηρίξει την ανταγωνιστικότητα και να υποστηρίξει την Ευρώπη εν γέννη. Ευχαριστώ την κυρία Μπιτζότο και τώρα η κυρία Ροντζούλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί Επίτροποι, θέτουμε το στόχο να δούμε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας για τα επόμενα χρόνια. Θέλουμε να δούμε το μέλλον των Ευρωπαίων νέων, των επαγγελμάτων, των οικονομιών που από αύριο θα υποστηρίξουν τις κοινότητές μας. Εδώ και αρκετό καιρό λέμε τι μορφέ εργασία θα έχουμε στα επόμενα 15 χρόνια, πώ θα αλλάξουν ε, οι δεξιότητε και τα προσόντα που απαιτούνται στην όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναρωτιόμαστε αν η παιδεία και η κατάρτιση που παρέχονται σήμερα θα χρησιμεύσουν στου νέου για να βρουν θέση εργασία. Αναρωτιέμαι πώ σκοπεύει η συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει τι νέε προκλήσει. Γνωρίζουμε όλε τι ανάγκε των νέων. Είμαστε βέβαιοι ότι το e-learning είναι η λύση ή θα πρέπει να μελετήσουμε νέε μορφές παιδεία και επιμόρφωση πιο συγκεκριμένε. Ε, Μα λείπουν μόνο έξι μήνε για να ολοκληρωθεί το πιλωτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε το Μάιο του 2010. Πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό. Θα έχουμε ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Θα πρέπει να εκπαιδεύουμε τους νέους με ευρωπαϊκές πολιτικές κατάρτισης που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες του μέλλοντος. Άκουσα ένα μεγάλο κατάλογο καθηκόντων, το τι πρέπει να κάνουμε, ε, να χρησιμοποιήσω και ιατρική ορολογία. Άκουσα πολλές διαγνώσεις αλλά καμία θεραπεία. Δεν θα πρέπει να ε, κάνουμε δημαγωγία, αλλά να βρούμε συγκεκριμένα μέτρα όπω απαιτεί η στρατηγική για το 2020. Αυτή είναι η πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη από κοινού με τι επιχειρήσει και αυτή είναι και η καλύτερη κληρονομιά που μπορούμε να αφήσουμε στα παιδιά μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Ροντζούλη. Η κυρία Εύελίνη Ρέγκνερ τώρα. μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, κυρία Επίτροπε. Νέε δεξιότητε, για νέε θέσει εργασίας. Είναι θέμα κλειδί αυτό, κομβικό, γιατί είναι για το μέλλον. Δεν πρόκειται μόνο ε, για τη δημογραφική ανάπτυξη, για την κρίση και πώς θα τα βγάλουμε πέρα πάνω κάτω μέχρι να περάσουν όλα αυτά. Όχι. Να δώσουμε τις ευκαιρίες των νέων με τα προσόντα και τις δεξιότητες να έχουν θέσεις εργασίας, να διαμορφώσουν το μέλλον για μια καινοτόμα οικονομία. Κύριε Επίτροπε, ε, ε, ποντάρετε πολύ στην συνεργασία των κοινωνικών εταίρων. Πολύ καλό αυτό. Τι γίνεται για τις συνθήκες εργασίας, για τα βαριά και τα αφηγηνά. Πόσο ε, επιβαρύνεται κάποιος και σωματικά και ψυχικά. Τι να το κάνουμε να έχουμε ε, τις καλύτερες επιδόσεις ε, από ένα εργαζόμενο σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και μετά μακροπρόθεσμα να καεί κυριολεκτικά και να μην μπορεί να αποδίδει. Δεν θα πρέπει ε, λοιπόν να λέμε μόνο για καλύτερη ρύθμιση, better regulation. Για το flexicurity λυπάμαι για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για να έχουμε ε, συμβάσεις ε, πρώτης εργασίας, εισόδου στην αγορά εργασίας. Δεν είναι καλό αυτό, δεν είναι πάρα πολύ φτηνό ε, να το επιφυλάσσουμε στους νέους που είναι το μέλλον μας το ίδιο. Από την αρχή, από την πρώτη θέση εργασίας να τους καταπιέζουμε τόσο πολύ και να τους υποβιβάζουμε μήπως ε, ομολογεί ότι βγαίνει νόκαουτ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παραδίδεται σε αυτές τις επισφαλείς θέσεις Παρακαλώ αυτό να το βελτιώσετε. Ευχαριστώ κυρία Γιούτα Στάινρουκ για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, κυρία Επίτροπε, πραγματικά η καταπολέμηση της ανεργίας είναι στόχος ε, μας και στόχος πλήρης απασχόλησης και είναι επίγον καθήκον. Το είπαν και άλλοι. Ο κόσμος στην Ευρώπη δεν θέλει έννοιες αόριστες και περιγραφέ, θέλει συγκεκριμένε λύσει. Ωραία αυτά που είπατε και οι δύο συνάδελφοί μου από την πολιτική μου ομάδα τα ανέφεραν, οι προλαλήσασε, αλλά ε, περισσότερη ευελιξία και περισσότερη κινητικότητα δεν δημιουργεί ούτε μία νέα θέση απασχόληση. Και θα ήθελα να τονίσω αυτά που είπε και η κυρία Σρόντερ και συμφωνώ. Χρειαζόμαστε θέσει απασχόληση, καλέ και ασφαλεί στην Ευρώπη και να φροντίσουν τα κράτη-μέλη και οι επιχειρήσει ότι είναι αορίστου χρόνου ε, και να μπορεί ο κόσμος να ζει από τα χρήματα που παίρνει. Αυτό να ξαναγίνει ο κανόνας και από την Ευρώπη να βοηθήσουμε και να δώσουμε και τα ορόσημα. Στην ατζέντα σας μιλάτε για νέες μορφές συμβάσεων εργασίας που επιδεινώνουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και μάλιστα στην πρώτη εργασία. Ε, εσείς τα λέτε ε, civil open contracts, αλλά αυτό δεν δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης. Πριν από μερικά χρόνια, όταν κυβερνούσε το κόμμα μου στη Γερμανία, το διαπίστωσε ε, τα ίδια τα μάτια. Δεν δημιουργούνται θέσει απασχόληση με την αποδυνάμωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Απλώ έχουμε μία μεταβίβαση ε, και μία μετάβαση από ε, σωστέ και ασφαλεί θέσει εργασία σε επισφαλεί και κακέ. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στη διαδικασία ΚΑΤΣΔΙ. Η πρώτη ομιλήτρια η κυρία Έλενα Μπασέσκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή είναι πολύ επίκαιρη. Δεδομένου ότι είναι αρκετά εθραστή ακόμη η ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας και τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν ε, δεινές συνθήκες στην αγορά εργασίας τους. Γι' αυτό και καλό θα ήταν η ευρωπαϊκή κοινωνία να στηρίζεται στη γνώση. Επίσης, ε, θα πρέπει να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς στην αγορά εργασίας. Και καλό είναι το εργατικό δυναμικό να έχει τα εφόδια και τις δεξιότητες για να μπορέσει να στελεχώσει τις νέες θέσεις εργασίας. Στη Ρουμανία είχαμε μια σταθεραποίηση της αγοράς εργασίας από τις αρχές του 2010. Δεν ε, νιώθουμε ακόμη όμως την ανάκαμψη, ούτε αντικατοπτρίζεται αυτή στη μείωση της ανεργίας. Δυστυχώς η νεολαία είναι από τις ε, πιο έθρευστες κατηγορίες και πάνω από 20% έχουμε ενεργεία των νέων. Είναι το πιο ευάλωτο με το πληθυσμό. Χαίρομαι για το στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αυξηθεί η απασχόληση στους νέους. Η κυρία Καταρίνα Ντάλοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν μιλούμε για ανεργία, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε την ανεργία των νέων, που είναι σχεδόν διπλάσια, για να μην πω μερικές φορές τριπλάσια από την ανεργία στα κράτη-μέλη. Καλή ατζέντα, αλλά δεν μας αρκεί μια απλή στρατηγική. Χρειαζόμαστε έμπρακτη εφαρμογή των μέτρων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να εκπονήσουμε και μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την αγορά εργασίας και τις απαιτήσει που θα έχει. Θα πρέπει να είμαστε πιο διορατικοί, να μην περιοριστούμε μόνο σε μια κοντόφθεμη στρατηγική, αλλά να δούμε τι θα, ποιες θα είναι απαιτήσει στο μέλλον από τους εργαζόμενους ή αυτούς που αναζητούν μια θέση εργασίας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε μια ανταγωνιστική οικονομία και ανταγωνιστική κοινοτικού Δεν θα πρέπει να περικόψουμε τους κοινοτικού προϋπολογισμούς, αλλά θα πρέπει να τους ενισχύσουμε γιατί οποιαδήποτε επένδυση στην παιδεία και την κατάρτιση θα είναι προσοδοφόρα. Παρακαλώ οι ομιλητές να μην μιλούν πάρα πολύ γρήγορα, διότι δυσκολεύεται τους ηρεμηνείς. Φραντς Obermeier. Ναι, ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στο κέντρο των μέτρων θα πρέπει να είναι ε, η βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντί να ποντάρουμε στη μαζική μετανάστευση, θέλουμε νέα προσόντα, η φόρα προσόντα βιώσιμα που να είναι προσαρμοσμένα στην οικονομία. Μετεκπαίδευση χρειάζονται οι πολίτες, εκείνοι που έχουν καταλήψει το σχολείο, την άσκηση ή το πανεπιστήμιο. Επίσης χρειάζονται κίνητρα για διαβίου μάθηση, για μετεκπαίδευση και κατάρτιση. Ειδικά για το 2011 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει μέτρα σε ε, κράτη-μέλη που ε, πλήττονται ιδιαίτερα από τη διάνοιξη της αγοράς και για εκείνους που έχουν χαμηλά προσόντα αλλά και για τους αυτοαπασχολούμενους που πέφτουν τα πρώτα θύματα σε αυτό το βωμό. Ε, καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το κοιτάξει αυτό και να τους προστατεύσει και από το κοινωνικό ντάμπινγκ αλλά και από τη φτώχεια τους ανθρώπους αυτούς. Ευχαριστώ. No. Ο κύριος Γιακολίνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε και κύριε Επίτροπε. Αδιαφεσβήτητα σε μια στιγμή τόσο μεγάλη δυσκολία για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δύσκολο να προχωρήσετε μια πρωτοβουλία σαν αυτή που παρουσίασαν οι Επίτροποι. Πρέπει λοιπόν να το δούμε με ευνοϊκό πνεύμα. Ε, παιδεία και κατάρτιση που στοχεύει να αποκτήσουμε δεξιότητες και γνώσεις που θα είναι χρήσιμες στην αγορά εργασία. Οι νέοι μέσω της ε, μόρφωσής τους και της κατάρτισής τους ε, θα πρέπει να εμπλουτίζουν συνεχώς τις γνώσεις τους. Έχουμε μια αγορά που χρειάζεται νέε δεξιότητε, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όσο δυνατόν περισσότερο τα μεταναστευτικά ρεύματα. Καλή αυτή οι τέσσερις στόχοι, αλλά θα πρέπει να λειτουργήσουν καλύτερα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα που είναι πολλά και τα έχει στη διάθεσή τη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τα νέα σύνορα της τεχνολογίας που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτές τις επιλογές, ώστε η στρατηγική του 2020 να συνάδει με την ε, ε, προσεκτική κατάρτιση και τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε μια αγορά εργασία που θα είναι στην υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως στην υπηρεσία των νέων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Finally, Η κυρία Τσικάου. Thank you very much, Mr. President. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η πρωταρχική ανησυχία των ε, Ευρωπαίων πολιτών είναι να διαφυλάξουν τη δουλειά τους Δυστυχώς ε, το ποστό ενεργείας ε, έχει φτάσει στα 10% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των ε, νέων μέχρι και 20%. Είναι πολύ δύσκολο να βρει κάποιο πια μια αγορά εργασία, ιδιαίτερα όταν είναι νέο και πολλέ φορές αρκείται σε πολύ επισφαλεί θέσει εργασία ή σε θέσει που είναι πολύ κατώτερες των προσόντων του. Η ατζέντα για τι νέε δεξιότητε θα πρέπει να συνδυαστεί με μια καλύτερη βιομηχανική πολιτική και πολιτική καινοτομία. Θα πρέπει να αναπτύξουμε το δυναμικό καινοτομία προκειμένου να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα και την ποιότητα των θέσεων απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, μια φιλοπεριβαλλοντική οικονομία στηρίζεται και σε νέε δεξιότητε. Εδώ θα πρέπει να ξεχνούμε και το θέμα τη πρόορη εγκατάλειψη των σπουδών. Πολλοί καταλείπουν τι σπουδέ ήδη από το Λύκειο. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη παιδεία στου νέου και να διευκολύνουμε την πρόσβασή του στην παιδεία. Τέλος, ο Επίτροπο Άντορ, εκ μέρου Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χαίρομαι ιδιαίτερος που ενστερνίζεστε τις ε, πρωταρχικές ε, ε, γραμμές αυτής της κοινωτικής πρωτοβουλίας για την πρόθεση της απασχολησιμότητας και την υλοποίηση ενός φιλόδοξου στόχου μέχρι το 2020. Φυσικά είμαστε σε φάση που θα περάσουμε από τη γενική συζήτηση στην επεξεργασία των λεπτομεριών αυτής της πρωτοβουλίας. Θα αναφερθώ σε ορισμένες παρατηρήσεις και σε μερικές κριτικές που ακούστηκαν. Καταρχήν, εμένουμε στην αρχή του flexicurity, της ευελιξίας με ασφάλεια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα δώσουμε έμφαση μόνο στην ευελιξία. Θα χρησιμοποιήσουμε ε, το flexicurity με κάπως διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Θα σας δώσω ορισμένα παραδείγματα όπου φαίνεται ότι λαμβάνουμε υπόψη τις νέες προκλήσεις και τους ε, καιρούς που διανύουμε. Ο ορισμός του flexicurity θα δίνει έμφαση και στην διαβιοκατάρτιση, γιατί είναι σημαντικές αυτές οι ευκαιρίες της διαβιοκατάρτισης και θα πρέπει να εξασφαλιστούν σε όλους τους εργαζόμενους. Γιατί πλέον ε, ο, η παραμονή στην αγορά εργασία ε, παρατείνεται. Γι' αυτό θα πρέπει να βοηθήσουμε περισσότερο τους εργαζόμενους με ευκαιρίες ε, αλλαγή στη σταδιοδρομία και με περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης. Καλό θα ήταν να δώσουμε έμφαση και στις δεξιότητες των νέων. Οι νέοι βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής του 2020, αλλά υπάρχει και ειδική πρωτοβουλία για τους νέους, η πρωτοβουλία νεολαία σε κίνηση. Και οι περισσότερες κοινοτικές στρατηγικές ε, λαμβάνουν υπόψη και τη σημασία των ε, νέων και η διάσταση νεολαία ε, είναι πολύ συγκεκριμένη στις περισσότερες πολιτικές δεν θέλουμε να ενισχύσουμε το flexicurity για τους νέους, γιατί ήδη είναι αρκετή και μάλιστα υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία για τους νέους εργαζομένους στην Ευρώπη από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Θέλουμε να διευκολύνουμε την κινητικότητα των νέων, γιατί πιστεύουμε ότι η νέα γενιά είναι αυτή που μπορεί να εκμεταλλευτεί καλύτερα την ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και να αναπτύξει τις σωστές δεξιότητες προκειμένου να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα αξιοποιώντας και τα νέα χαρακτηριστικά της αγοράς αλλά και τις δυνατότητες ε, και τους θεσμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μίλησα προηγουμένως για καλύτερες συνθήκες εργασίας και για ποιοτικές θέσεις απασχόλησης. Λυπούμε που δεν το κατάλαβε αυτό η κυρία Σρέτερ. Η κυρία Σρέτερ και είπα ότι ο κατακαιρματισμός της αγοράς εργασίας είναι σημαντική πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και μάλιστα αναφέρθηκα σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, τα open-ended contracts, τις ανοιχτές συμβάσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποτρέπουμε τη σύναψη συμβάσεων αορίστη μόνιμων συμβάσεων, απλώς θέλουμε να βοηθήσουμε όσους μέχρι στιγμής είχαν μόνο συμβάσεις περιορισμένου χρόνου εργασίας, ορισμένου χρόνου εργασίας, τους δίνουμε την ευκαιρία να έχουν ανοιχτέ συμβάσεις αορίστου. Νομίζω ότι αυτό σε κάποιο βαθμό θα βελτιώσει όχι μόνο τις θέσεις απασχόλησης, αλλά τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και αυτό είναι σημαντικό όταν μιλούμε για ποιοτικέ θέσεις εργασίας. Και όταν μιλούμε για επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, στο ανθρώπινο κεφάλαιο, δεν θα πρέπει να αμελούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υποστηρίζει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες σε όλα τα κράτη-μέλη. Και ευελπιστούμε ότι το ΕΚΤ θα παραμείνει ένα εύρωστο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα στηρίζει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Πρόκειται για δεκαετίες πρωτοβουλίες που θα ισχύσουν για όλα τα κράτη-μέλη. Δεν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε άμεσες ε, ε, οικονομικές ανάγκες των κρατών μελών ή κατεπίγουσες ε, περιστάσεις. Έχουμε έναν δεκαετή ορίζοντα διορατικό δηλαδή και δεν είναι μια πολιτική που θα αντιμετωπίζει τις κατεπίγουσες περιστάσει. Φυσικά η στρατηγική αυτή θα ισχύσει και για την Ελλάδα και για την Ιρλανδία. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που θα μπορούσε να βοηθηθεί από μεγαλύτερη ευελιξία για να βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα, όπως και η Ισπανία. Και η Ιρλανδία είναι μια χώρα που θα μπορούσε να επανισορροπήσει τους παράγοντες της ανταγωνιστικότητας και να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην επένδυση των δεξιοτήτων και της επιμόρφωσης σε σχέση με άλλες πηγές ανταγωνιστικότητας που μέχρι στιγμής χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερο στην τελευταία περίοδο στην Ιρλανδία. Και φυσικά να ε, δοθεί έμφαση στην κρίσιμη κατάσταση που αντιμετωπίζουν ε, οι χώρες αυτές και μέχρι του χρόνου μάλλον δύσκολα θα αν, αναβαθμιστεί το επίπεδο της απασχολησιμότητας αλλά θα πρέπει να έχουμε μια γενική εικόνα και επισκόπηση. Πιστεύω ότι από το δεύτερο εξάμεινο του επόμενου έτους αρχίσει η βελτίωση της κατάστασης γιατί οι μεγαλύτερες οικονομίες ε, ήδη έχουν παρατηρήσει μια αύξηση των θέσεων εργασία, ήδη αρχίζουν και βιώνουν την ανάκαμψη και παρά τι διαφορέ και τι δυσκολίε στο χρηματοπιστωτικό τομέα ε, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία και θα εφαρμοστούν οι ευρωπαϊκέ πολιτικέ. Και μπορεί η μικροδιαχείριση να μην γίνει δυνατή από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη-μέλη, αλλά θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τι πρωτοβουλίε μα για όσο δυνατό μεγαλύτερη απασχολησιμότητα. Τέλο τη συζήτηση, σα ευχαριστώ πολύ και περνάμε τώρα στι ερωτήσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο, κύριος, Επίτροπος Άντορ είναι ο πρώτος ε, επίτροπος που θα απαντήσει όταν είναι έτοιμος μπορεί να απαντήσεις στην ερώτηση 17 του κυρίου